Ωραία. Έληξε αυτή η συζήτηση και όπως γνωρίζετε θα ψηφίσουμε αύριο στις 11.30 την έκθεση αυτή και τις τροπολογίες της. Θα ήθελα να σας κάνω ορισμένες ανακοινώσεις. Καταρχήν να σας πω ότι λάβαμε από το Συμβούλιο δύο θέσεις για πρώτη ανάγνωση που θα πρέπει να εγκρίνουμε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής. Οι τίτλοι θα παρουσιαστούν στην ε, παρούσα Ολομέλεια, στην παρούσα Σύνοδο. Και η διαδικασία ξεκινάει από τις 26 Οκτωβρίου. Από τους πράσινους έλαβα ένα αίτημα διορισμού που ε, εντάσσεται στην παρούσα σύνοδο και εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρούμε ότι εγκρίνεται ο εν λόγω διορισμός ή διορισμοί. Το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η διορισμη το επομενο θεμα Γκάρδια Θάμπαλ Ρουμπιάλ για τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα μέσα στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το λόγο έχει ο κύριος Καρδιαθάμπαλ, ο εισηγητής. Η κυρία μάλλον. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος λέει ο πρόεδρος. Ε, για τρίτη φορά παρεμβαίνω στην Ολομέλεια και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις και τους γνωμοδότες. Υπάρχουν τρεις